βεβαίω ότι οι ανησυχίε σα σε αυτό το τομέα ε, είναι και ανησυχία τη Κομισιόν και αφορούν τον τομέα τη έρευνα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προβλέπονται έτοιμα ε, πρώτα ψηφίσματος των Φιλευθέρων, των Πρασίνων, των, ε, της Γκουε και των Σελιστών. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο το μεσημέρι στις 11.30. Ολοκληρώθηκε έτσι για το θέμα τη ημερήσια διάταξη και έτσι πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσια διάταξή μα, τι παρεμβάσει διαρκείας ενός λεπτού δυνάμει το άρθρο 150 του κανονισμού μας με πρώτο ομιλητή το κύριο Σκυλακάκη. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως με την Αίγυπτο. Πρέπει στο δύσκολο επόμενο διάστημα να ενεργοποιηθεί στο μέγιστο η εξωτερική υπηρεσία για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών στην Αίγυπτο, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αίγυπτο, αλλά και των ιστορικών θεσμών που τις εκπροσωπούν όπως το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Στο βασικό μου θέμα τώρα, τα απορρίμματα. Ενώ έχουμε ένα υψηλού επίπεδου νομοθετικό πλαίσιο όλα σχεδόν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαδικασίες επί παραβάση. σε πολλά αναφέρονται κρίσεις σκουπιδιών και υπάρχουν τομείς όπου καταγράφεται μαζική παραβίαση του κοινοτικού δικαίου όπως οι διασυνοριακές μεταφορές απορριμμάτων. ταυτόχρονα τα κράτη μέλη για λόγους πολιτικούς το περίφημο όχι στη δική μου αυλή δεν συμμετέχουν όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε στην προσπάθεια χρειάζεται λοιπόν η επιτροπή να προτείνει νέα συμπληρωματικά εργαλεία όπως η επέκταση των αρμοδιοτήτων του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και η δυνατότητα αποστολών της ένωσης για εξακρίβωση στοιχείων στα κράτη μέλη. Ας τα σκεφτεί αυτά η Επιτροπή εν ώψη των προτάσεων του 2012. Ευχαριστώ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην κατάσταση στη Ρουμανία γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου. Κύριος Νικολέσκου, μέλος της αντιπολίτευσης, συνελήφθηκε. Αυτό ανακοινώθηκε πριν ε, να υλοποιηθεί. Ανακοινώθηκε η σύλληψη πριν να γίνει έτσι. Λοιπόν, να καταλαβαίνετε ότι η εξουσία δεν λειτουργεί δημοκρατικά, δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης οδηγούν ε, στο να βγαίνει ο κόσμος στο δρόμο και μιλάμε για πολίτε οι οποίοι είναι φτωχοί. Εγώ θέλω να ευστήσω την προσοχή σας σε όλα αυτά. Η κυβέρνηση επίσης αγόρασε εξοπλισμό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, για να σκίσει καταστολή στον κόσμο. Πρόκειται για πολιτική δικτατορία στη Ρουμανία και αν δεν ληφθούν κυρώσει τώρα τι θα γίνει. Στο μέλλον εμείς ε, διαμαρτυρόμαστε κατά αυτών των πολιτικών κατακρίσεων. Ζητάμε εμεί ω Ένωση ε, το σεβασμό τη δημοκρατία στην Τινησία, στην Αίγυπτο, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμό δημοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Τα προβλήματα των καπνοπαραγωγών στη Βουλγαρία, λέει ο κύριο Μετίν Καζάν, ε, γεννούν πολλές δυσκολίες σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Και συλλαλητήρια διαμαρτυρία, στο οποίο συμμετέχουν δεκάδε χιλιάδων πολιτών που διαμαρτύρονται για την κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για την παραγωγή καπνού. 17 είναι οι χώρες οι οποίες παράγουν καπνό και όλες αυτές στηρίζουν τους παραγωγούς τους με επιδοτήσεις. Όμως η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα όπου δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα, αυτή η επιδότηση. 76 εκατομμύρια ευρώ είχε είχαν σχεδιαστεί για να στηρίξουν τον καπναπαραγωγό της Βουλγαρίας, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια του. Κύριε σήμερα σε ένα αξιοσημείωτο κλίμα ομοφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε την έκκληση του Προέδρου του κυρίου Μπούζεκ για να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμως τη γενοκτονία των Ρωμά ε, που ήταν θύματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί. Είπε μάλιστα ότι οι Ρωμά αποτελούν μια μειονότητα την πιο καταπιεσμένη για μακρύ χρονικό διάστημα. Σε ποιους απευθυνόμαστε όμως, ποιο θα εφαρμόσει τι πολιτικέ που συναποφασίζουμε. η κομισιόν είχε παραγγείλει από τον ιούλιο του 2008 μια έκθεση για τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για του ρωμά που αφορά 18 χώρε την οποία έχει στα χέρια τη ήδη από τον ιούνιο. έκανα λοιπόν σχετική ερώτηση γιατί ε, θεωρώ ότι είναι απολύτω αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στην δημοσιοποίηση μια τέτοια πολύτιμη έκθεση. έγινε και διεθνή κίνηση δημοσιοποίηση η κυρία ρέντινγκ απάντησε στην ερώτηση και δεσμεύτηκε στη δημοσιοποίηση μέχρι το τέλος του δεκεμβρίου του. 2010. ήδη έχουμε φεβρουάριο και η έκθεση δεν δημοσιοποιήθηκε. θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω το γιατί. Ο κύριο Τζόκο, ξέρω ότι δεν ήταν σωστή η προφορά μου. Ζόμπρο, ζόμπρο. Αλλά εντάξει, σας κατάλαβα, λέει ο κύριο Ζόμπρο. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις σε σχέση με την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος και άλλων βλαπτικών αερίων. Τα μέτρα τα οποία λύθησαν κατά αυτών των συζητήσεων, λέγω, ήταν πάρα πολύ ζημιογόνα για τις επιχειρήσεις και για με την κατάσταση πολλών ε, βιομηχανιών που φύγανε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σας λέω ότι τα όσα είπαμε δεν ελήφθησαν υπόψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να, μάθαμε ότι για από τη Γερμανία, την Πολωνία, βιομηχανίες τώρα ε, πασχίζουν το πώς θα μετεγκατασταθούν να πάνε στην ΕΣΔ ή στην Νότια Αμερική. Θα πρέπει να ληφθεί δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επομένω ε, βλέπουμε να υπάρχει κανένα όραμα σχετικά με αυτό. Η κυρία οραμα σχεδον η κυρια φικερεντο και πραγματικά σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ θέλω να διαβάσω, όπως ε, υποσχέθηκα και στους πολίτες, ότι το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, οργάνωσε την περασμένη εβδομάδα ε, μια κραυγή που ένωσαν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις για την καταπολέμηση της κρίνης και για τις μεγάλες επιπτώσεις που υπάρχουν στην ανεργία, στην κοινωνική ανισότητα και στη φτώχεια. Παρά το 2010 ήταν το έτος κατά της φτώχειας. Εκεί ζητήθηκε οι δραστηριότητε και οι εργασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντικατοπτρίζουν την οργή των οργανώσεων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της στόχης λαμβάνοντας υπόψη την ε, κρίση και τις συνέπειές της, ε, ο κοινωνικός απακλισμός και η φτώχεια ε, αναφέρονται σε διάφορες προτάσεις αλλά πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταγγείλει την κατάσταση αυτή δημιουργώντας μια ομάδα εργασίας που ε, θα αναλάβει να αναλύσει τις κρίσεις στον κοινωνικό τομέα και να μελετήσει τα μέτρα που θα... Επόμενος ομιλητής παρακαλώ, κυρία Φιγκερέντο, όχι δεν γίνεται. Σας παρακάλεσα, δεν μπορείτε να ξεπεράσετε το ένα λεπτό. Αυτό επιβάλλει ο κανονισμός. Πρέπει να ρίχνουμε και μια ματιά στο ρολό Είχαμε μακρά ημερήσια διάταξη σήμερα και πολλή δουλειά. Και γι' αυτό τώρα παρακαλώ τον κύριο Μαρινέσκου να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγκρίναμε αυτές τις, αυτά τα μέτρα για τη Ρουμανία και Καταλήξαμε στο ότι όλα τα σχετικά με το Σέγγεν τα πληρεί. Η Ρουμανία όμως δεν μας αφήνουν να μελετήσουμε αυτά τα έγγραφα οπότε πώς τα ψηφίσουμε. Τα είπε αυτά η Επιτροπή των ε, Δημοκρατικών Ελευθεριών. Ζητήσαμε τον αποχαρακτηρισμό αυτών των εγγράφων και όπως έχω το σήμερα τα πράγματα νομίζω ότι δικαιούται η Ρουμανία να υποβάλει στο Κοινοβούλιο όλες τις σχετικές εκθέσεις προσχώρησης ή στο Σέγγεν. Νομίζω ότι μόνο με αυτές τις εκθέσεις είναι δυνατόν να ληφθεί η σχετική απόφαση. Εάν δεν υπάρχουν και άλλου είδους κριτήρια, αυτό αντιβαίνει στις ε, ιδρυτικές συνθήκες, στο κοινωτικό δίκαιο, γιατί έκανε ό,τι επέτασε ο νόμος η Ρουμανία όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Επομένως θα πρέπει να λάβει την απάντηση που της αξίζει. Ευχαριστώ κυρία έχει το λόγο τώρα. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η δημοκρατία στη Ρουμανία ποτέ δεν υπέστη πιέσει όσε τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε ήδη κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τη στάση του Προέδρου της, ε, ε της Κάτω Βουλής, ο οποίος παραβιάσει κάθε έννοια ε, κράτους δικαίου και αποδεικνύεται με τις τελευταίες εξελίξεις ότι το κυβερνητικό κόμμα, το κυβερνών κόμμα στη Ρουμανία έχει στο στόχαστρο τις ελευθερίες, τις πολιτικές και τα δικαιώματα των πολιτών. Το Δημοκρατικό Φιλελεύθερο Κόμμα έχει κηρύξει τον πόλεμο σε ολόκληρο τον ρουμανικό λαό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα δημοκρατικό μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντιδημοκρατικό, να ε, συλλαμβάνει αυθαίρετα και να τιμωρεί για λόγους βεντέτας όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο στην, σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Χάκη, έχει το λόγο τώρα. Κυρία Πρόεδρε, ω ε, ευρωβουλευτή από την Ιρλανδία, ζητώ να λάβετε υπόψη την αδύνατη οικονομική κατάσταση στην Ιρλανδία. Ναι, υπάρχουν πολλέ αποτυχίε, αλλά δεν ε, τα πράξαμε μόνοι μα. Ε, Επενδύσει πάρα πολλέ χώρε εισέρευσαν στι Ιρλανδικέ τράπεζε και κατέρευσαν σε χαρτίν πύργη και τώρα οι Ιρλανδοί φορολογούμενοι πληρώνουν, το άθο πληρώνουμε 5,8% σε τόκους και μα έχει επιβληθεί δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα λιτότητα 4 ετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί αυξάνεται η ανεργία, αυξάνεται η μετανάστευση και για τέταρτο έτος έχει μειωθεί το ΕΠ και όπω και η ΕΚΤ δίνει 132 δισεκατομμύρια και τα αφήνει στην προστινή πόρτα των ελληνικών τραπεζών 110 ε, δισεκατομμύρια έφυγαν από την πίσω πόρτα το 2010 ε, από την πίσω πόρτα των τραπεζών. Έτσι λοιπόν πολύ, γρήγορα η κατάσταση γίνεται μη βιώσιμη και όπως είπε ο κ. Ε, η Ευρώπη ε, είναι τμήμα της λύσης και χρειάζεται να ληφθεί σοβαρή δράση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντότ έχει το λόγο τώρα. Ε, Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα μόνο στη δική μου εκλογική περιφέρεια της Βόρειας Ιρλανδίας τοποθετήθηκαν στο βόρειο Μπέλφαστ δύο βόμβες και μόνο ο Θεός μας έσωσε και δεν μιλάμε σήμερα για εκατόμβι νεκρών. Μπορούσαν οι δυνάμεις ασφαλείας να σώσουν εκατοντάδες πολιτών που ε, εκένωσαν την περιοχή πολύ γρήγορα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια σειρά από δολοφονικές επιθέσεις εις βάρος αστυνομικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας. Και ξέρω Πρόεδρε ότι δεν ενδιαφέρουν τα μέσα ενημέρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά Μα υπενθυμίζουν αυτές οι τρομοκρατικέ ενέργειες ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μα φέρουν στο ζωφερό δρόμο της τρομοκρατίας. Και όταν πριν τα Χριστούγεννα ο κύριο Μπαρόσο σε συνάντηση με τον κύριο Ρόμπινσον επιβεβαίωνε τα καθήκοντα της ομάδας Μπαρόσο, εγώ χαιρέτησα αυτή την προσπάθεια και την στήριξη τη συνευτικής διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ είχαμε όλα αυτά τα σχόλια τα αρνητικά τα σχετικά με την Ουγγρική Προεδρία όμως τα βέλη δεν ήταν κατά το προγράμματος της Προεδρίας τα βέλη αυτά εστράφησαν κατά τις νομοθεσίες για τα ΜΜΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ήδη πει τις απόψεις της προς την κυβέρνηση και η κυβέρνηση είπε ότι θα αναθεωρήσει τη τάσεις της, θα τροποποιήσει αυτή την νομοθεσία αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε το ίδιο όσον αφορά ε, γίνεται νομοθεσία στη Σλοβακία για τη γλώσσα που ακόμα ισχύει και ακόμα ε, επιβάλλουν χρηματικές κυρώσεις σε κόσμο που χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα. Αυτοί μας που καίγονται για το δικό μας νομικό τα γιατί δεν αγανάκτησαν και αυτά τα οποία ε, επευλήθησαν κατά της ουγγρικής μηνότητας στη Σλοβακία. Πολλοί τράχτηκαν πάρα πολύ από εκείνο το χαλί στο Συμβούλιο από έναν παλιό χάρτη της Ουγγαρίας. Μα πρόκειται περί συμβόλου. Περί συμβόλου το οποίο θα βοηθούσε μια ισχυρή Ευρώπη εάν ε, αξιοποιούσαμε και εκτιμούσαμε τις αξίες της Κύριε Πρόεδρε, στις 14 Φεβρουαρίου έχουμε τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο οποίος και αυτός είχε υποφέρει από επιληψία, γι' αυτό είναι η μέρα επιληψίας. 39.000 στη Σκωτία υποφέρουν. 20.000 επίση έχουν διαγνωστεί, λαμβάνουν φάρμακα και επομένω έχουμε όλου αυτού οι οποίοι κάθε μέρα κινδυνεύουν να πάθουν κάποια κρίση και αν το προβάλλουμε αυτό σε όλη την Ευρώπη σημαίνει ότι εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη ζουν με αυτό το φόβο. Στι 14 Δευτέρα επομένω θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και θα πρέπει να καλύψουμε όλου αυτού που του έχει διαγνωστεί ασθένεια, ε, να βοηθηθούν από ειδικού νευρολόγους για την επιληψία στις 15 Φεβρουαρίου θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις στο Κοινοβούλιο και παρακαλώ συνάδελφοι ελάτε θα έρθει και κόσμος από την εκλογική περιφέρεια και με την ευκαιρία να ε, χαιρετήσω δύο ειδικού από την Σκωτία οι οποίοι πρόκειται να παραστούν. Ευχαριστώ κύριο Ζέδη, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να ε, μιλήσω για το εξής. Μου είπαν ε, πρόσφατα ε, ότι δεν υποστηρίζουν τα ΣΕΚΕΛ. Όμως ε, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, έχουν δικαίωμα στην αυτονομία και στην αυτοδιάθεση. Θέλω να σας ε, ενημερώσω ότι η αυτοδιάθεση είναι μια, ένα δικαίωμα που είναι διεθνώς αποδεκτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει σε ορισμένες μειονότητες τη δυνατότητα να έχουν αυτονομία, ενώ κάποιε άλλε όχι, δηλαδή οι Βάσκοι ναι, ε, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι λοιπόν, ε, αν δεν υποστηρίζετε ε, την αυτονομία αυτών των ανθρώπων, τότε δεν σέβεστε τι αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Σκέλη έχει το λόγο. Πρόεδρε, τι θέλω να πω ότι η ελευθερία διακίνησης εργασίας είναι, μια, ε, ένας από τους κύριους στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ε, ελευθερία εργασίας δεν υπάρχει. Ένα ταλός, αν θέλει να δουλέψει στη Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει να περιμένει 9 μήνες για να πάρει άδεια. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της αναγνώρισης ε, των δεξιοτήτων, ειδικά αν θέλουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ηλεκτρονικής υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νοσέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάχρηση της ε, εξουσίας ε, ε, στο οποίο προβαίνει η κυβέρνηση της Ρουμανίας σημαίνει ότι βρίσκεται από το 1989 σε μια πολύ σκοτεινή στιγμή ε, η κυβέρνηση της Ρουμανίας ε, το στέχμα παραβιάζεται θεωρητικά υπάρχει διάκριση των εξουσιών αλλά μια και μόνο εξουσία ο πρόεδρος ελέγχει τα πάντα και κάνει ό,τι θέλει καθημερινά προβαίνει σε κατάχρηση της εξουσίας θέλει να καταστρέψει την αντιπολίτευση και να φημώσει οποιαδήποτε αντίθετη φωνή που προτείνει εναλλακτική στην κυβέρνησή του. Δεν πρέπει να παραμείνουμε αδιάφοροι σε αυτά που συμβαίνουν στη Ρουμανία, ε, ούτε εδώ ούτε στα υπόλοιπα κρατημέλη. Όλοι θα πρέπει ε, να αποκαλύψουμε τι συμβαίνει και ούτε πρέπει να παραπλανηθούμε από τις εξηγήσει ε, των ε, κυβερνώντων στη Ρουμανία ή από τους συμμάχους τους. Τα γεγονότα αρκούν ε, για να δούμε την πραγματικότητα στη χώρα μου που είναι θλιβερή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιβαν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα Παρεμπιπτόντω να υπενθυμίσω τον πρόεδρό μα κάτι σε σχέση με την εξέλιξη δημοκρατία στην Ρουμανία. Διότι ο πρόεδρο είχε βρεθεί στη χώρα και στήριξε την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι ανίσχυρο ουσιαστικά το κοινοβούλιο στην χώρα μα. Η κυβέρνηση περνάει του νόμου. Αλλά με τις Ελλάδες και εκείνη δεν έχει πάρα καμία ιδιαίτερη εξουσία γιατί ο πρόεδρος της χώρας τους διορίζει τους υπουργούς. Αυτός αποφασίζει για τα μέτρα που λαμβάνονται οπότε μπαίνουν οι ένοχοι στη φυλαϊκή ένα μήνα και κατόπιν περνάνε από δίκη. Επίσης κάτι άλλο για τον πρόεδρο Μπουζέ Θα πρέπει να υπάρξει μια τοποθέτηση επίσημη και να υπάρξει κατόπιν απάντηση επίσημη του πρόεδρου Μπασέσκου. Ακόμα περιμένω να το κάνει αυτό ο κύριος Μπούζεκ. Ο κύριος Μίρσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τι νομίζετε ότι ε, εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν υιοθετεί τα ψηφίματά του. Υποθέτω ότι τα υιοθετεί προκειμένου να εφαρμόζονται. Πλην όμω φαίνεται ότι η λετωνική κυβέρνηση σκοπεύει να υιοθετήσει, να εφαρμόσει μάλλον ε, το ψήφισμα τη 11η Μαρτίου του 2004, το οποίο ξεκάθαρα ορίζει ότι η Λετωνία θα πρέπει να χορηγήσει το δικαίωμα της ψήφου στις ε, δημοτικές εκλογές σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της Λετωνίας. Πότε σκοπεύει η Λετωνία να ε, εφαρμόσει αυτήν την ε, διάταξη ε, στα αγγλικά λέμε όταν αρχίσουν να πετάνε τα γουρούνια, στα ε, λετωνικά λέμε όταν ε, ανθίσει ο παλιός τάβλος, στα ρωσικά λέμε όταν αρχίζουν να σφυρίζουν οι σολομοί. Ε, αυτό λοιπόν θα είναι και η εποχή που θα μπορέσουν να ψηφίσουν οι ρωσόφωνοι κάτοικοι της Λετωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έντσου. Danke schön, asistăm Εμείς ε, είδαμε κάποια γεγονότα που θα αλλάξουν την ιστορία της Βορειάς Αφρικής ε, και όχι μόνο τα δικτατορικά καθεστώτα δεν μπορούν να συνεχίσουν στην εξουσία. Θέλω να βυστήσω την προσοχή σας ε, στο ότι υπάρχουν μορφές διδακτατορίας και σε ένα κράτος βόλος που θεωρείται δημοκρατικό τη Ρουμανία. Μιλάμε πάντα για το τεκμήριο της αθωότητας. Ε, πάντοτε πρέπει να κρίνεται κάποιος ε, χωρίς να έχει προφυλακιστεί αν δεν αποτελεί δημόσιο κίνδυνο όμως ε, αυτό δεν ισχύει ε, για τον πρόεδρο Μπατσέσκου και για τους υπόλοιπους που είναι στην εξουσία η δήλωση του κυρίου Μπατσέσκου στο Στρασβούργο πριν πέντε μήνες ε, πριν από την σύλληψη του Κωνσταντίνου Κολέσκου είπε ότι ένα σημαντικό μέλος της αντιπολίτευσης συνελήφθη και μάλιστα ούτε καν είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο ε, αυτό ο άνθρωπος ε, τι περισσότερο χρειάζεστε για να καταλάβετε πώς ασκεί την εξουσία ο κύριος Μπασέσκου. Ευχαριστώ κυρία Κρέτσου, έχει το λόγο. Δεν έχετε ανάψει το μικρόφωνο σας κύριε Κρέτσου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στη δίωξη της αντιπολίτευσης στη Ρουμανία. Κάθε φορά η κυβέρνηση ασκεί όλο ένα ε, και μεγαλύτερη αυθαιρεσία ε, το ιδιωτικό επίπεδο είναι πολύ κακό και η κυβέρνηση λαμβάνει όλο ένα και πιο αντιδημοκρατικά μέτρα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Όπως ε, είπε και ο συναδελφό μου, ένα από τα μέλη τη αντιπολίτευση συνελήφθη. Αυτό ε, μα δείχνει πώς απειλείται η αντιπολίτευση και ταυτόχρονα ο εθνικό προπολογισμό χρησιμοποιείται για του πελάτε τη κυβέρνηση, Τα μέτρα της ε, κυβέρνησης οδήγησαν σε κοινωνικέ διαμαρτυρίε και εμεί συμφωνούμε με τι διαμαρτυρίε αυτέ, έναντι των όσων κάνει η κυβέρνηση κατά τη αντιπολίτευση και των συνδικάτων πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα κατά της παραβίασης των δικαιωμάτων στη Ρουμανία. Και τελευταίο έχει το λόγο ο κύριος Κόρτες Λάστρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία τα πούμε για αυτό το ένα λεπτάκι, αλλά όμω θα πρέπει σε αυτό το λεπτό να σα πούμε κάτι που μα ικανοποίησε, διότι πρόσφατα υπογράφηκε ένα κοινωνικό συμβόλαιο στην Ισπανία μεταξύ των συνδικαλιστών, τη κυβέρνηση και των επιχειρηματιών. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία την αναδεικνύει την Ισπανία ω χώρα η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιε δυσκολίε και τι ε, ε, προκλήσει αυτέ και να προχωρήσει στο κράτο ε, τη ευημερία και πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση και προσδίδεται επομένω ευθύνη σε όλη την κοινωνία. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα κερδίσουμε την πρόκληση για το μέλλον και πώ θα οικοδομήσουμε μια δυνατή Ισπανία σε μια ένωση πρωταγωνιστή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ολοκληρώνουμε δηλαδή την ημερήσια διάταξη για τη σημερινή συνεδρίαση αύριο, 5η, 3 Φεβρουαρίου 2011. Έχουμε συνεδρίαση από τις 9 μέχρι, τις, μέχρι τη 1